ευθούν αυτές οι νομικές πράξεις στα πρακτικά της παρούσας ε, συνόδου. Κατόπιν η κυρία Πάσκαλ Γκρινή με ενημέρωσε γραπτός ε, ότι εκπνέει η θητεία της ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι εξελέγει στην Γαλλική Βουλή. Βάσει του άρθρου λοιπόν 7 παράγραφος 2 όπου ε, προβλέπονται διατάξεις περί εκλογών και βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1 και 4 του κανονισμού, του ιστορικού κανονισμού, αποφασίζουμε ότι χειρεύει πλέον η έδρα της από 14 Δεκεμβρίου 2010 και μετά κατόπιν. Η ομάδα ε, των Δημοκρατών και Φιλελευθέρων μου ζήτησε